Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πάρα πολλοί έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο στο πλαίσιο των επεξηγήσεων ψήφου. Ε, αλλά το αργότερο που μπορούμε να τελειώσουμε είναι 3 παρατέταρτο για να μπορούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμάσουν την αίθουσα για τη συνεδρίαση στις 3 ε, η ώρα. Ε, και όσοι δεν μπορέσουν να λάβουν το λόγο σήμερα, ίσως μπορούν να το λάβουν αύριο μετά την ψηφορία και οι υπόλοιποι μπορούν βέβαια να καταθέσουν και τις επεξηγήσεις τους σε γραπτή μορφή. Ο κύριος Κόρμπετ για ένα λεπτό. ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενώ συζητούσαμε αυτό το θέμα χτες, ο κύριος Φαράζ έθεσε ένα ζήτημα που καμία σχέση δεν είχε με την έκθεση και αφορά όμως ε, το θέμα που έχει να κάνει με την προστασία του λαβρακιού. Ε, και μετά ε, με αυτή την αφορμή άρχισε να επιτίθεται κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επειδή εγώ είμαι πολλά χρόνια εδώ μέλος, ξέρω περίπου πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση, δεν την έκανε μάλλον οι υπουργοί των κρατών μελών έλαβαν την απόφαση με την οποία διαφωνούσε συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Τζότζιού ε, σα, που είναι ο Βρετανός συντηρητικός υπουργός. Αντί να στρέφει τα πειρά του όμως τους υπευθύνους για την απόφαση, τη ίδια στρεβλώνει και τη στρέφει κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό τι δείχνει είτε αγνία είτε κινησμό και προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει αυτό ως θέμα στο ερχόμενο Βρετανικό δημοψήφισμα. Αυτά τα πράγματα είναι ε, τελείως ιδεχθή και επονίδιστα. Τόρες ε, Μαρτίνες. Joder, no me va esto, no me enciende. No. ¿Sí? Puedes hablar. Μπορείτε να μιλήσετε, λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Ναι, ευχαριστώ. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να μιλήσει με τόση φασαρία και τόσο λίγο σεβασμό προ του ανθρώπου που μιλάνε αυτή τη στιγμή σε επεξηγής ψήφου. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να τονίσω το εξή. Παρά το γεγονό ότι αναβλήθηκε η έγκριση, ε, της έκθεσης έχει βελτιωθεί ε, το στόκ και το απόθεμα του ερυθροπτέρυγου τόνου αλλά δεν ακολουθεί η ποσόστοση. Οι αλλοί μα τα λένε αυτά, κάνουν πολύ σκληρή δουλειά κάθε μέρα και εδώ εμεί ψηφίζουμε το μέλλον και τι ζωέ των ανθρώπων. Ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ε, μοιράζει ε, στην Ισπανία τις ποσοστώσεις. Μιλούμε για τον ερυθροπτέρυγο τόνο, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη τόνου και άλλα αλλιεύματα που κάθε μέρα χάνονται. Όπως είναι η παλαμίδα, ας πούμε, εκείνη που εξαφάνιση. Δεν είναι λοιπόν έντιμα όλα αυτά. Η κυριαρχία είναι κάτι το οποίο ορισμένοι καταχρώνται και εις βάρος των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση αυτή εμείς θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχε καμία ε, τεκμηριωμένη ε, μελέτη της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των αλλιευτικών κοινοτήτων. Και γι' αυτό τη βρίσκαμε έτσι κι αλλιώς επονίδιστη. Ε, δεν ψηφίστηκε η έκθεση, επαναπέμφθηκε στην Επιτροπή για να την ξαναμελετήσουν. Χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά οι αλληλείς και στη Μεσόγειο και στις ε, Κανάριες νήσους, στον Ατλαντικό, θα πρέπει να ανακτήσουν την ποσότητα που δικαιωματικά τους αναλογεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαμίκινς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι το σχέδιο ψηφίσματος έχει στόχο να βελτιώσει την πραγματική εφαρμογή της ε, κοινή αλευτικής πολιτικής ε, για ε, τον τόνο στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό ωκεανό. Υπάρχουν παραδοσιακές αλευτικές κοινότητες που χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους ε, και αλλιευτικά εργαλεία. Αυτοί αντιμετωπίζουν ε, τεράστιες δυσκολίες. Δεν θα πρέπει να απειλούμε εμείς με τις ενέργειές μας και τις αποφάσεις μας ε, τις κοινότητες αυτές. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η επιβίωση των αλλιέων. Ένα άλλο θέμα είναι οι απορρίψεις των ειδών που ε, αλλιεύονται παραπλεύρως. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ κύριο Χάνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει βεβαίως νόημα το να κρίνει κανείς μια οργάνωση με βάση τα πεπραγμένα της. Ε, είχαμε εδώ τον πρόεδρο της Επιτροπής που ήρθε και μας είπε πώς πρέπει να επεκταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια κοινή πολιτική για τα φορολογικά και άλλα. Άρα δηλαδή το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι πώς ακριβώ τα πήγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τομείς που ήδη υπάρχει νομοθεσία. Η κοινή ελευτική πολιτική εισήχθη το 1972. Ας δούμε λοιπόν λιγάκι το ιστορικό, ε, να δούμε ε, πώς έχουν χειριστεί τα αποθέματα στη Βόρειο Θάλασσα. Βλέπουμε ε, το τι συμβαίνει στην έκθεση που κατατέθηκε και βλέπουμε ότι υπάρχει οικολογική καταστροφή, έχει ε, καταστραφεί μια ανανεώσιμη πηγή. Υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα πρέπει να τους βάλουμε να εποπτεύουν το στρατό ή οτιδήποτε άλλο. το, λόγο έχει ο κύριος Γούλφ. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα ένας και μόνο επίτροπος από τη Μάλτα εισάγει ένα κανονισμό, όχι μια οδηγία, ένα κανονισμό που θα επηρεάσει 800.000 ε, αλληλείς ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο που ψάχνουν τα ψάρια και τώρα ένας άνθρωπος ε, που δεν τον έχει εκλέξει κανείς στην Ευρώπη τους λέει ότι θα μπορούν όλοι να ψαρεύουν μόνο από ένα ψάρι. Και αυτό ε, δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε με την εξουσία των λαών. Μόνο με το τι πιστεύει η ελίτ ότι είναι σωστό κάποτε ελέγχτη κανείς δεν είναι αρκετά καλός για να ε, κυβερνά χωρίς τη συνένεση των υπολείπων. Αν αυτό το καταλάβαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η διακυβέρνηση είναι από το λαό, για το λαό και αυτό πάλι το έχει πει κάποιος άλλος μεγάλος ότι η εξουσία δεν είναι για τους ίδιους ε, που την κατέχουν. Ε, πρόεδρος, για να διευκρινίσω κάτι, σήμερα το Κοινοβούλιο ψήφισε. Ο κανονισμός κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σήμερα ψήφισε το Κοινοβούλιο. Ε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν μιλώ να έχετε καλοσύνη να με ακούτε, γιατί αλλιώς και εγώ τι νόημα έχει να σας τα λέω αυτά που σας λέω. Έχετε την καλοσύνη να με ακούτε. Κοιτάξτε, εγώ ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα ψήφισε το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ψήφισε αυτόν τον κανονισμό. Οι κανονισμοί δεν επιβάλλονται από τους επιτρόπους, αλλά ψηφίζονται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Άρα δηλαδή υπάρχει σύνομοθέτηση, δεν υπάρχει αυταρχική επιβολή. Απλά ήθελα να το διευκρινίσω. Τώρα πάμε στο επόμενο στις εκθέσεις ε, Λάγκε και Κόρμπιτ. Ο κύριος Κόρμπετ έχει το λόγο. Η έκθεση αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πραγματών της πολιτικής ανταγωνισμού με την ευρύτατη έννοια. Και υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια που είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτή τη στιγμή το οποίο έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει η χαλιβουργία μας με ένα dumping από τους ε, Κινέζους χαλιβοπαραγωγούς. Αυτό είναι θέμα ανταγωνισμού αλλά και θέμα εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και καιρό έχει ε, προτείνει να ενισχύσουμε την άμυνά μας σε τέτοιες περιπτώσεις και Υπάρχει μια χώρα που τα καθυστερεί όλα αυτά, που δεν μας αφήνει να παίρνουμε αποφάσεις. Και ποια είναι αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βρετανική συντηρητική κυβέρνηση είναι ένας από τους υπετίους και τους ενόχους για την κατάσταση αυτή και δεν μας βοηθάει, δεν ενισχύει την κατάστασή μας να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία. θα μπορούσαν να είχαν αναλάβει εθνική δράση, γιατί το προβλέπει η συνθήκη αυτό στα άρθρα για τον ανταγωνισμό, δεν το έπραξαν και ορισμένοι μπαίνουν στον πειρασμό καμιά φορά να κάνουν αυτό που πάντα κάνουν και είναι πάγια τακτική να τα ρίχνουν όλα στις Βρυξέλλες. Σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που έχουν ζητήσει το λόγο για επεξήγηση ψήφου και δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά τις 3 τέταρτο. Γιατί μετά στις 3 ξαναρχίζει η ολομέλεια. Σας παρακαλώ να σέβεστε τους χρόνους, γιατί όσο εσείς μιλάτε περισσότερο, τόσο λιγότερο μιλητέ θα μιλήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και σεβασμό προς τους συναδέλφους μας. Θα δώσω μέσα το λόγο στην κυρία Μόρβαη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή, πρέπει να σας πω, ε, ότι μου άρεσε ιδιαίτερα το σημείο σε ορισμένε μετακομμουνιστικές χώρες έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε για να προστατεύουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία, διότι αποτρέπει τη συγκέντρωση οικονομικής εξουσίας και πολιτικής στα χέρια των ολίγων. Διότι ε, αντιτάσσεται σε κάποιες φεουδαρχικές δομές που ακόμα κρατούν τα ενία της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά χρήματα και μοιράζουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια στους ε, αριστούς τους. Αυτά όλα είναι σημεία που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και όταν έχουμε πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα σύστημα με ίσους κανόνες παιχνιδιού προς όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως φιλίας. Ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πολιτική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια από τις πιο αποφασιστικές αρμοδιότητες της Ένωσης και επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη. Ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην διεθνή σκηνή. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία όμως ανάμεσα στα συμφέροντα των καταναλωτών από τη μία και στις ανάγκες για ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων από την άλλη. Αυτός είναι ένας από τους στόχους της συγκεκριμένης έκθεσης. Αν έχουμε ανάγκη λοιπόν την κοινωνική συνοχή και για να γίνει αυτό χρειάζεται βελτίωση των εθνικών πολιτικών και στον τομέα των φορολογικών τους δραστηριοτήτων και της αντιμετώπισης των μονοπωλιακών ή μονοπωλιακών καταστάσεων. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση, πρέπει να τα υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο, έτσι θα προστατεύσουμε την διεθνή ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεών μας. Η κυρία Μακοβέη. Εγώ ψήφισα διαφορετικά από την πολιτική ομάδα. Νομίζω ότι μια υγιής μορφή του φορολογικού ανταγωνισμού είναι αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, την φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους που κοστίζουν σε ετήσια βάση, λέει η ομιλήτρια, χίλια δις. Λοιπόν, βλέπουμε ότι από την άλλη υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν τους φόρους τους και κάποιες άλλες οι οποίες ε, διαφεύγουν. Πρέπει να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις να μην προσφεύγουν στους φορολογικούς παραδείσους και να πληρώνουν τους φόρους τους εκεί όπου έχουν ε, βγάλει τα κέρδη τους. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την έδρα τους ε, στους φορολογικούς παραδείσους δεν μπορεί να συμμετέχουν στους διεθνείς διαγωνισμούς. Έτσι θα βοηθήσουμε την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κέλλη. Θα να πω ε, ελπίζαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε θέσεις απασχόλησης και να δημιουργήσουμε και νέες θέσεις απασχόλησης. Θέλω λοιπόν να πω μερικά πράγματα για ορισμένες από τις ε, τροπολογίες. Ε, ούτε εγώ, ούτε οι συνάδελφοί μου ψηφίσαμε όπως ψήφισε η ομάδα μας στις τροπολογίες 76 και 89 παραδείγματος χάρη. Εκεί δηλώσαμε αποχή γιατί ε, συνδυάζουμε το CCTB και εμεί δεν συμφωνούμε επ' αυτού. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα μόνο των κρατών μελών, τα φορολογικά δηλαδή. Επιπρόσθετα απήχαμε στην τροπολογία 81-2 ε, γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεπερνάει και την πρωτοβουλία ECCPPS. Ε, σας λέω υπάρχουν πάρα πολλές καλές συστάσεις. Ε, χαιρετίζει κυρίως αυτά που λέγονται για τους αγρότες και για τις ε, τιμές ε, που επιτυγχάνουν. Αυτό βέβαια κάπως πρέπει να αλλάξει το μέλλον. Χάναν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από το 30% έχει πέσει το ΑΕΠ του συνολικά στο 17% το 15%. Και πού οφείλεται δεν λέω ότι αυτό οφείλεται μόνο στο ότι αναπτύσσονται οι αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν υπάρχει κάτι παραμπερές ούτε στη Βόρεια Αμερική ούτε οπουδήποτε αλλού. Γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι υπερβολικές ρυθμίσεις και δεν μιλάω μόνο ε, για τη REACH και άλλες οδηγίες, η MFID παραδείγματος χάρη που καταστρέφουν ε, τις θέσεις απασχόλησης, αλλά μιλάω και γι' αυτό το λόμπι ε, το οποίο θέλει να υπάρχουν κανόνες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ευνοούνται οι μεγάλες τράπεζες και να ε, στριμώχνονται οι μικροί ανταγωνιστές. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ πολλές επιχειρήσεις αν θέλουν να επιτύχουν αναγκάζονται να φύγουν από την Ένωση. Όσο λοιπόν παραμένει στη ζωή αυτό το σύστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταδικασμένη να συνεχίσει να βαίνει την κατιούσα. Ε, Μαγκίνες παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία η έκθεση αυτή και ιδιαίτερα στις παραγράφους 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 σαν γνωμοδότρια για τις εμπορικές αθέμητες πρακτικές στην αλυσίδα εμπορίας τροφίμων. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε προτάσεις έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό των αθέμητων πρακτικών και νομίζω ότι θα πρέπει τέτοιου είδους ιδέες να ενταχθούν στο έγγραφο αυτό. Εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή. Ταυτόχρονα συμφωνώ ότι οι νομοθέτες έχουν καθήκον να προωθούν ένα οικονομικό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό όμως πρέπει να βοηθά τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις νέες αγορές και να αποσύρει τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στις εμπορικές δραστηριότητες. Uh, Υπάρχει έρευνα για συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες στη Βόρεια Ιρλανδία σε σχέση με την πιθανή δημιουργία δραστηριοτήτων λόμπι. Η απόφαση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναδρομική ίσπραξη σε σχέση με τις έρευνες για το σχιστολιθικό αέριο είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στις μικρές αυτές εξορικτικές επιχειρήσεις και μάλιστα όταν δεν πρόκειται για κάποιο λάθος το οποίο είναι δική τους ευθύνη θα πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση αυτή και μπορέσουν να λειτουργήσουν καλή την πίστη οι εξοριστικές αυτές δραστηριότητε. Η κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή για την πολιτική ανταγωνισμού περιλαμβάνει πάρα πολύ θετικέ προτάσεις. Μεταξύ αυτών το θέμα των κρατικών ενισχύσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα που μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στον κλάδο. Εγώ συμφωνώ με τα όσα λέγει η έκθεση ότι θα πρέπει να αναλυφθεί κάποια μέρημνα έτσι ώστε να μην καταστραφεί ε, ή στρεβλωθεί ε, ο ανταγωνισμός υπέρ των μεγάλων τραπεζών. Στην Ιρλανδία από τις αρχές ε, του χρόνου υπάρχει περιορισμός στις καταθέσεις που μπορεί κανείς να έχει σε ένα ταμιευτήριο. 100.000 ευρώ. Αυτά δεν είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει πρόβλημα και θα πεταχθούν εκτός της ε, ε, κτηματαγοράς ε, αυτοί οι οργανισμοί. Αυτό είναι κατά του ανταγωνισμού και ένας τέτοιος κανονισμός δεν συνάδει με την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι υπέρ της δεσμευτικής δράσης στις επιχειρήσεις, τα σούπερ μάρκετ που ταλαιπωρούν καταναλωτέ και αγρότες. Ο Μίλτον Φρίμα, λέει ο κύριο Κούβουλφ, είπε κάποτε ότι οι τέχνες ε, ε, γνώρισαν πρόοδο ε, όχι από κεντρικέ κυβερνήσεις και πάρτε όποια τέχνη θέλετε. Εδώ που βρισκόμαστε το επίκεντρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η συγκεντρωτική διαχείριση ε, στο Συμβούλιο και από μη εκλεγμένε επιτροπέ. Και εδώ στον ανταγωνισμό και τη συγκεκριμένη πολιτική για άλλη μια φορά βλέπουμε πως αυτή η συγκεντρωτική κυβέρνηση θέλει να ελέγξει τι ε, επιχειρήσει και πώ το πράττει. Έχουμε συγκεντρώσει τα νομίσματά μας στο ευρώ και βλέπουμε τη ζημιά στην ευρωζώνη και, ποια, και πόση ανεργία για τους νέους είναι αυτό. Οι κεντρικοί κανόνες και οι κανονισμοί τι δείχνουν και πώς επιδρούν ε, στο εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα πρέπει λοιπόν να εξαγάγουμε εμεί ω δίδαγμα εδώ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει πια να συγκεντρώνεται, να επιστρέψει στα εθνικά κράτη και να είναι ελεύθερη για να ανταγωνίζεται παγκοσμίω στους υπολείπους. Περνάμε τώρα στην έκθεση Word. Κυρία Μόρβαη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο διαπολιτισμικός διάλογος ε, είναι το αντικείμενο της έκθεσης αυτής και δυστυχώς δεν μπόρεσα να την υπερψηφίσω, διότι δεν κάνει λόγο για αξίες, για αρχές, για θέματα μιλάει για διάφορα θέματα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Μα πώς μιλάς για διαπολιτισμικό διάλογο όταν βλέπεις γυναίκες στην Ευρώπη να βγαίνουν στο δρόμο την παραμονή της πρωτοχρονιάς για να γιορτάσουν τον ερχομό του νέου έτους και να υφίστανται επιθέσεις. Αυτά δεν τα συζητάμε στο διαπολιτισμικό μας διάλογο, δεν μας απασχολούν. Μπορούν οι Ευρωπαίες να ταξιδεύουν με το τρένο χωρίς να συνοδεύονται από άρενα. Είναι ζήτημα αυτό στην Ευρώπη. Μπορεί μια Ευρωπαία να πάει μόνη της σε μια πισίνα και να μην κινδυνεύει. Αυτά δεν τα συζητάμε στο διαπολιτισμικό διάλογο. Δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα, δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην ισότητα. Και όσοι τα αμφισβητούν ανήκουν είτε στη φυλακή είτε πίσω στις χώρες τους από όπου μας κουβαλήθηκαν. Μίτσι. Όταν κάποιος σχολίασε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιστορία της, είπε ότι θα είχε ξεκινήσει από την παιδεία και τον πολιτισμό. Οι επόμενες γενιές για να γίνουν υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας πρέπει να σέβονται τη διαφορετικότητα και να καταπολεμούν τις διακρίσεις, τη βία, την ριζοσπαστικοποίηση και την ξενοφοβία. Συγχαίρω λοιπόν την εισηγήτρια και υπεψήφισα την πρότασή της. Βλέπω με ευχαρίστηση ότι και η δική μου πρόταση είχε γίνει δεκτή. Πρέπει να εκτίθενται τα παιδιά σε άλλους πολιτισμούς από μικρή ηλικία για να αναπτύσσουν τις σωστές αντιλήψεις. Αυτό θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, την ευρωπαϊκή και την έβρεση θέσεων απασχόλησης. Νομίζω λοιπόν ότι οι σχολικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι στραμμένες και προς άλλες χώρες έτσι ώστε στα παιδιά από μικρή ηλικία να μπορούν να εκτιμήσουν την διαφορετικότητα των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών. Έτσι θα δημιουργήσουμε τους αυριανούς ηγέτες ένα, μια κοινή αίσθηση του ανήκειν στις ευρωπαϊκές αξίες. Ο κύριος Μαμίκης. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτισμική ποικιλομορφία έχει σχέση με τον διαπολιτισμικό διάλογο, με την αμοιβαία κατανόηση, γιατί η εκπαίδευση είναι καθοριστική σημασίας στην κοινωνία μας. Δεν μπορεί να γνωριθεί πουθενά στον κόσμο. Γιατί υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό να στηρίξουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου τη διαφύλαξη της ε, πολιτισμικής ε, ταυτότητας ε, σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό, είναι και καθοριστική σημασία. Επίσης είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε όλες αυτές τις αρχές έχοντας κατά νου το μέλλον και διασφαλίζοντας ε, την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ο διαπολιτισμικός διάλογος, διάλογος μεταξύ πολιτισμών είναι κάτι που έχουμε ζήσει στην Ευρώπη ανέκαθεν. Δεν είναι ένα καινοφανές φαινόμενο με το τελευταίο κύμα της μετανάστευσης. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικότητες για λόγους ιστορικούς και λοιπούς. Έχουμε κοινότητες που συμβιούν. Ο δια... πολιτισμικός διάλογος δεν έχει σημασία μόνο σε σχέση με τη μετανάστευση και με τη σημερινή διάσταση, αλλά είναι πολύ σημαντικός για να ε, καλύπτονται και οι ανάγκες κάποιων αυτοχθόνων μειονοτήτων. Αυτή η έκθεση λοιπόν το τονίζει αυτό είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης, ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι προς όφελος όλων και δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν το έχουν προσέξει πάρα πολύ αυτό. Υπάρχουν θεμητά αιτήματα και καθόλου αδικαιολογημένα αυτοχθόνων μειονοτήτων και κοινοτήτων. Ο διαπολιτισμικός διάλογος δεν λειτουργεί πάντα στα κράτη-μέλη, γι' αυτό στρέφονται ε, οι μειονότητες αυτές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσουν τη βοήθειά της. Ελπίζουμε να ε, είναι πιο ευήκον το ους των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στο μέλλον. Η κυρία Πετήρ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ την έκθεση αυτή την υποστήριξα πρέπει να σας πω διότι ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος είναι αποφασιστική για την κατανόηση των ανθρώπων. Έχουμε ποικιλομορφία και θα πρέπει αυτή να γίνεται σεβαστή. Δυστυχώς σήμερα χωλαίνει αυτός ο διάλογος και στην Ευρώπη καμιά φορά λησμονούμε που θεμελιώσαμε τις κοινωνίες μας ε, και που εδράζονται και ε, ε, οι αξίες και οι αρχές μας. Γι' αυτό στα πλαίσια του διαλόγου αυτό θα πρέπει να τονίζουμε και το ρόλο της οικογένειας, διότι κυρίως εκεί μαθαίνει κανείς ε, τον ίδιο του το πολιτισμό, στο κύτταρο της οικογένειας που αποτελεί τη βάση της ίδιας μας της κοινωνίας και εμεί θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύουμε την οικογένεια και τις αξίες με τις οποίες γαλουχούμε τα παιδιά μας. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την οικογένεια, ή μάλλον εάν διατηρήσουμε την οικογένεια και τη διαφυλάξουμε, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τον πολιτισμό μας. Γιατί αν μεγαλώνουμε σωστά τα παιδιά μας, τότε θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Κύριος Πόλτσακ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ την υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι ο πολιτισμός και η μόρφωση μας βοηθούν για να κατανοούμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Αυτά όλα τα λέει το άρθρο 5 άλλωστε τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αξίε όπω είναι το κράτο δικαίου. Γι' αυτό οι αξίε αυτέ θα πρέπει να προστατεύονται και να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζουμε και εκείνε τι κοινωνίε που δεν το έχουν καταλάβει, δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει ο διαπολιτισμικός διάλογο να είναι κάτι διαφορετικό από την πολυπολιτισμικότητα. Προσοχή, υπάρχουν κίνδυνοι εδώ δεν θα πρέπει να απεμπολίσουμε την ταυτότητά μας και τις ρίζες μας και να τις φέρνουμε στο ίδιο επίπεδο με την πολιτισμικότητα. Υπάρχουν χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα οι κοινωνίες τόσο πολύ ώστε να τα κατανοούν όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία Ντότς. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι μέλος του Κοινοβουλίου από τη Βόρεια Ιρλανδία και αναγνωρίζω πλήρως με τα σχηματισμό που μπορεί να γίνει στο μυαλό νέων ανθρώπων ε, όταν ε, έχουν θετικές εμπειρίες από ανθρώπους που έρχονται από άλλο κόσμο, έχουν άλλες πεπιθήσεις. Και ξέρω πόσο επικίνδυνη είναι η ριζοσπαστικοποίηση. Είδαμε στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες τι έγινε. Υποστηρίζω πλήρως όλα εκείνα τα μέτρα που θα βοηθήσουν να σταματήσει η στρατολόγηση νέων και ε, που υποστηρίζουν το τερματισμό του διχασμού και της διχόνοια. Θα πρέπει να στείλουμε τα σωστά μηνύματα παντού στην Ευρώπη, αλλά έχει σημασία εδώ στη μάχη αυτή ε, να έχουν τον πρωταγωνιστικό σημαντικό ρόλο οι κυβερνήσει των κρατών μελών. Η έκθεση προσπαθεί να επηρεάσει το ρόλο της εθνικής πεδίας προσπαθεί να εναρμονίσει την νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά και την πολιτιστική έκφραση. Αυτά τα θέματα είναι θέματα κυριάρχων κυβερνήσεων να τα αποφασίζουν και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν έχουμε διχόνια επιτόπου σε μια κοινότητα, από εκεί θα πρέπει να προκύπτουν οι λύσει. Και οι αμετανόητοι φεντεραλιστέ, σήμερα εδώ θα πρέπει να τα καταλαβαίνουν αυτά και να τα ακούνε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην έκθεση Μπάλ σε Μορβάη παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ δεν υπερψήφισα αυτό τον κανονισμό περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διότι γίνεται λόγος για όλα αυτά ε, που θα γίνουν στο μέλλον, που όμως ε, ήδη έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν και είναι πολύ σημαντικό να, ε, να προσέξουμε λίγο το θέμα των ενυπόθηκων δανείων πρέπει να δίδονται σωστές ε, πληροφορίες σε ανθρώπους ε, που ομιλούν ε, για τις τράπεζες να έχουμε κατά νου την σωστή τραπεζική εποπτεία. Αυτό το θέμα το έθιξα στον Επίτροπο, δηλαδή ρώτησα τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει όλους εκείνους που δεν είναι σε θέση ε, να, πληρώσουν τα, να αποπληρώσουν τα ενώπικα δάνειά του. Μαμίκινς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα πλαίσια της ε, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης προκλήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα διαρθρωτικού τύπου που εξακολουθούν να ε, χαρακτηρίζουν σήμερα τις αγορές κεφαλαίων όπως επίσης και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίε. Ο ρόλος μας ως νομοθετών δεν έχει εξαντληθεί. Όλα τα θεσμικά όργανα τα οποία έχουν λόγο σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να εφαρμοστούν ε, νέα μέτρα μεταρρυθμιστικά και αποτροπής μελλοντικών κρίσεων. Ένα από τα μαθήματα που πήραμε το 2007-2008 ήταν η ανεπάρκεια εποπτείας και παρακολούθησης των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε υποχρεωτική τη λήψη κάποιων νομοθετικών μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δε εφαρμογή τους προσέκρουσε σε διάφορες δυσκολίες στα κράτη-μέλη. Επίσης, υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις αντιφατικές μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη έκθεση λοιπόν εξετάζει όλα αυτά τα κενά και τις ελλείψεις και προτείνει ε, μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τώρα την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου το οποίο προέκυψε από την κρίση και που ε, λίγο άρον-άρον συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πρέπει τώρα να έρθουμε να διορθώσουμε όλα τα στρεβλά που ε, αποφασίστηκαν τότε λόγω της ταχείας λήψης των αποφάσεων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη διαφάνεια ε, της υλοποίησης και της εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων. Είδαμε λοιπόν τα μέτρα που λάβαμε ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εκ τότε μεσολάβησαν πολλά χρόνια και είδαμε πώς η οικονομική κρίση εξελίχθηκε και τι κατεύθυνση πήρε. Και τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι απαρχαιωμένα και να χρειάζονται νέα. Καπούτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω επέμβει επανειλημμένα σχετικά με το θέμα των ε, νομοθετικών διατάξεων για τα χρηματοψηφιακά. Με αυτή την έκθεση ε, κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, ε, κυρίως όσον αφορά τα αριθμιστικά για τις χρηματοψηφιακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην ζήσουμε μια άλλη ύφεση όπως αυτή του 2008. Τώρα πλέον πολλοί μιλούν για μια επιδημία στην, ε, στον τομέα της ενέργειας, ε, κυρίως όσον αφορά σε σχέση με το σχιστολιτικό αέριο. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν ε, οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και εγώ συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι δεν υπάρχει ενιαία νομοθετική ρύθμιση αυτό αφορά όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους και ο στόχος μας είναι η χρηματοψηφιακή σταθερότητα, η προστασία των καταναλωτών και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των χρηματοψηφιακών τομέων που απειλείται από την Κίνα και από το Brexit, ε, από την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, αυτά ε, καθιστούν ότι ε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά τους κινδύνους. Κέλλη παρακαλώ. Ε, ήμουν εδώ ε, στην προηγούμενη θητεία και είδα όλες τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από εσάς ε, τότε ήταν επίτροπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και για να υπάρξει νομοθεσία που θα διασφαλίζει ότι δεν θα επανέλθουν αυτά τα προβλήματα. Καλό λοιπόν τώρα που κάνουμε απολογισμό για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σωστό ε, που κοιτάμε λίγο το μέλλον. Ο τελευταίος ομιλητής αναφέρθηκε στις ε, ενδεχόμενες συνέπειες ε, του σχιστολιτικού αερίου για τις εταιρείε και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Άρα δηλαδή πρέπει να επαγρυπνούμε εμείς χαιρετίζουμε την Τραπεζική Ένωση και την πειταρχία που θα επιφέρει στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Όπως αναφέρθηκε, πρέπει ε, να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολτσακ, παρακαλώ, επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα την έκθεση πρωτοβουλία στη συγκεκριμένη θεωρώ ότι δείχνει το είδος των προβλημάτων τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κεφαλογικών αγορών. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ξεκινούν τη δραστηριότητά τους και κυρίως τα προβλήματα χρηματοδότησής τους θα δούμε ότι το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ε, βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη και των υπηρεσιών και της επιχειρηματικότητας. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ε, αρνητικά και για τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την καινοτομία. Υποστηρίζω λοιπόν τις προτάσεις οι οποίες γίνονται και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περαιτέρω προτάσεις στον τομέα των κεφαλογικών αγορών. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Βαλίνα. Ναι, έκθεση κυρίας Ματέρα. Ευχαριστώ. Bien, las... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε ε, υποταγμένες στην κοινωνία, ούτε θα καθόμαστε να μας λένε τι πρέπει να κάνουμε. Πόσο μάλλον όταν κυριαρχούν οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις ει βάρο των πολιτών. Οι γυναίκες όπως και οι άντρε, έχουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε για το μέλλον μας, για το αν θέλουμε να είμαστε ε, μητέρες ή όχι παντρεμένες ε, ή ανήπαντρες, επιχειρηματίες ή εργαζόμενες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η οχι παντρεμενες η ανηπαντρε επιχειρηματιε η εργαζομενε σε καμια περιπτωση δεν αυτή που προτείνεται για να ε, σταματήσουν οι αδικίες προς τις γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθεί πολιτικές ε, κατά ε, της μισθολογικής διαφοράς και που να προωθούν ε, τη συμφιλίωση του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο. Να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες για να μπορούν οι γυναίκες να αναπτύσσονται απολύτως και με ανθρώπινο τρόπο και συνεργασία τους ό,τι και να θέλουν να κάνουν. Και όχι να τους δίνονται κίνητρα για να καλύπτονται οικονομικοί κλάδοι ανάλογα με τα τρέχοντα συμφέροντα της οικονομίας. Οι λιτότητες που επέβαλε η Ένωση και πολλά τελευταία χρόνια έπληξαν σφοδρά τις συνθήκες διαβίωσης πολλών πολιτών και οι γυναίκες ε, πραγματικά είναι εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο και από τη φτώχεια και από τη δουλειά και από την οικογένεια. Θα πρέπει διαπαντός να εγκαταληφθεί η ιδέα ότι η γυναίκα ε, με την υποταγή της ε, είναι κάτι που χρησιμοποιούμε εμβαλωματικά για να καλύπτουμε τις πληγές ε, ε, στην οικονομία. Όλα αυτά οφείλονται στην ανισότητα και το βλέπουμε καθημερινά. Άρα Βεβαίω να ενισχύσουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, βοήθεια για όποια γυναίκα πλήρη υποστήριξη, αλλά όχι εκμετάλλευση τη γυναίκα. Γι' αυτό η ομάδα μα ψήφισε αποχή. Σα ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εμεί πολύ. πολύ. Μιλήσατε εκ μέρου ε, τη ΓΚΟΕ, Κοράτσα Μπιλτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σα πω ότι στηρίζω ανεπιφύλακτα την έκθεση, γιατί η γυναική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα ε, μοναδικό δυναμικό για την ποιότητα για να αποκτήσει κανείς εξουσίες. Εμείς δεν είμαστε ευάλωτη ομάδα. Οι γυναίκες είναι σημαντικοί βασικά στοιχεία στην οικονομία μας αποτελούν κεφάλαιο της οικονομίας και έχει έρθει πια στιγμή τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν πλήρως ε, το δυναμικό αυτό της ελληνικής, ε, της ε, γυναικείας επιχειρηματικότητας. Να μην υπάρχουν διακρίσεις, να αρθούν τα εμπόδια και να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στο κεφάλαιο, να περιστεί η γραφειοκρατία, να μην υπάρχουν διακρίσεις, επίσης να αντιμετωπιστούν και τα στερότυπα. Πολλές φορές οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ω ε, ως περισσότερο ευάλωτες. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση, να υπάρχει ένας, μια ανατροπία της δεύτερης ευκαιρίας, έτσι ώστε οι γυναίκες να πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ε, χαιρετίζω λοιπόν ε, το ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα δίκτυα γυναικών. Είναι σημαντικό να αλληλοστηριζόμαστε, να μάθουμε μία από την άλλη. Επίσης τα κράτη-μέλη πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τις γυναίκες για να συνδυάσουν καλύτερα την εργασία με την οικογένειά τους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Τζιτνάνσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια για μια έκθεση που ε, αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις γυναίκες φυσικά, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, ε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς τα προβλήματα των γυναικών. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι γυναίκες ή για τον τρόπο με τον οποίο θα ανατρέψουν τα παιδιά τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο, περισσότερο χρόνο, μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας και καλύτερη σχολική ε, δραστηριότητα για τα παιδιά. Έτσι μόνο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες οι οποίες εργάζονται και οι οποίες κάποια στιγμή θα ήθελαν να γίνουν ε, ε, επιχειρηματίες. Κλούνε. Ε, υποστηρίζω με ευχαρίστηση τη συγκεκριμένη πρόταση για τη διευκόλυνση των γυναικών στον επιχειρηματικό χώρο. Νομίζω ότι συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα θέματα της ανεργίας στην Ευρώπη για να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ξεκινούν τη δραστηριότητά τους και έχουν πραγματικά τεράστιες δυνατότητες έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Εμπόδια στον τομέα της πρόσβασης σε ε, δανεισμό, σε ρευστότητα, αλλά και προβλήματα σε σχέση με τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ασχολούνται με τα παιδιά τους, φροντίζουν τα παιδιά τους. Και νομίζω ότι οι κυβερνήσεις είναι σε θέση να πάρουν μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τις γυναίκες επιχειρηματίες. Εμείς φυσικά θα πρέπει να αφήσουμε τις γυναίκες ελεύθερες να αποφασίσουν, αλλά κάποια θέματα όπως ο ευέλικτος χρόνος απασχόλησης πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η κυρία Μόρβάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι ε, επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αναφερθούμε στις γυναίκες και στις δυνατότητές τους γενικότερα, να δούμε τι εμπόδια αντιμετωπίζουν στις μετακομμουνιστικές χώρες, στη δική μου χώρα σαν παράδειγμα στην Ουγγαρία. Δεν υπάρχει δυνατότητα ρευστού για τις γυναίκες αυτές έτσι ώστε να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Έχουμε επίσης ε, και τα θέματα της ιδιωτικοποίησης των κομμουνιστικών αγαθών και κεφαλαίων. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους ε, έτσι ώστε να φύγουν σε δυτικές χώρες και τα χρήματα αυτά βρίσκονται στα χέρια των επενδυτών χωρίς να έχουν ξεκινήσει προγράμματα που θα επιτρέψουν να υπάρξει διαθέσιμο κεφάλαιο για τις ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπόρζον, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η γυναική ε, επιχειρηματικότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από πολύ αυξημένε δυνατότητε δανειοδότηση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν οι γυναίκε να δημιουργήσουν νέε επιχειρήσει. Ε, στην Κροατία έχουμε μάλιστα μια εθνική στρατηγική προκειμένου να προωθήσουμε τη γυναική επιχειρηματικότητα. Η έκθεση λοιπόν αυτή τη κυρία Ματέρα λέει ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντικέ οικονομικέ αλλαγέ αλλά και κοινωνικέ αλλαγέ. Επομένω την υποστηρίζουμε πλήρω. Ευχαριστούμε πολύ. Μάμικινς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόνο 31% ήταν γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλο δρόμο να διανύσουμε όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά και όσον αφορά και τη σωστή ισορροπία μεταξύ οικογενειακού βίου και εργασίας. Και εδώ βεβαίως εισφέρουν οι κοινωνικές ενισχύσεις, οικογενειακά επιδόματα κλπ. Πέραν τούτου ε, θα πρέπει να προωθήσουμε το ήθος της επιχειρήσης ιδιαιτέρως ε, σε τομείς όπου οι γυναίκες έχουν μια δυνατότητα εξέβρεσης εργασίας. Ούτως ώστε να υπάρχει σωστή ισορροπία το, και ούτως ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί μας το 2020, δηλαδή μια συμμετοχή στα 80% ε, στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από νομικής πλευράς ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διαφορετική νομική αντιμετώπιση όσον αφορά τους άνδρες και τις γυναίκες στο ζήτημα της επιχειρηματικότητα. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι ε, το 1 τρίτο των επιχειρηματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 1 τρίτο, είναι γυναίκες. Κύριε Επίτροπε, προφανώς χρειαζόμαστε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό, προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε πιο ισότιμες συνθήκες πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τελικά στην επιχειρηματικότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις συμμετοχής γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε ικανούς υποψηφίους για τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Προφανώς ε, οι διορισμοί θα πρέπει να γίνονται αξιοκρατικά. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε επαγγελματίε επιχειρηματίες Παρ' αυτά θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Ο κύριο Κέλλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά συζητάμε ένα ζήτημα το οποίο έχω παρακολουθήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οφείλω να σας πω ότι όταν πρωτοείδα τα αριθμητικά δεδομένα σε σχέση με τους άνδρες και τις γυναίκες επιχειρηματίες, μου προξένησε εντύπωση η πολύ μεγάλη απόκληση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα και αναρωτήθηκα για ποιο λόγο μια τέτοια διαφορά. Ένας από τους σημαντικούς λόγους θεωρώ ότι είναι η ίδια η αυτοπεποίθηση. Ζήτημα το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο και στα δύο φύλλα και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην περίπτωση των γυναικών προκειμένου και οι γυναίκες να έχουν αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και να μπορούν και αυτές να γίνουν εξίσου επιχειρηματίες με του άνδρες, να έχουν τι ίδιε δηλαδή ευκαιρίε. Α μην ξεχνάμε όμω επίση ότι πολύ συχνά ορισμένοι πιστεύουν ότι οι γυναίκε επιχειρηματίε δεν έχουν τι ίδιε δυνατότητε δανειοδότηση, χρηματοδότηση, ίδρυση ε, επιχειρήσεων. Βλέπω σιγά σιγά κάποιε αλλαγέ όμω και στην ίδια μου τη χώρα, την Ιρλανδία. Δημιουργούνται νέε επενδυτικέ πλατφόρμες που προωθούν τι ε, επενδυτικέ επενδύσει των γυναικών. Νομίζω ότι τέτοιε εθνικέ προσπάθειε θα πρέπει να ενθαρρυνθούν. Πετήρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο των ε, γυναικών ε, επιχειρηματιών στη χώρα μου είναι μόνο 13%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 23% που είναι γυναίκες επιχειρηματίες και ένα πολύ μικρό ποσοστό γυναικών που όμως είναι ιδιοκτήτες των ίδιων των επιχειρήσεών τους. Τα πράγματα διαφέρουν πολύ βέβαια από τα δεδομένα που είχαμε το 2001, όταν μόνο 7% των γυναικών στην Κροατία ήταν επιχειρηματίες. Υπάρχει όμω ένα τεράστιο περιθώριο βελτίωση ακόμα. Όπω βλέπουμε και στην έκθεση αυτή, υπάρχουν πάρα πολλοί εξωτερικοί παράγοντε που αποτελούν εμπόδιο στη γυναική επιχειρηματικότητα, ιδίω όταν προσπαθούν να δημιουργήσουν νεοφυεί επιχειρήσει, start-up κτλ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δημιουργήσουμε εμεί τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό άχθο που βαρύνει τι γυναίκε επιχειρηματίε και να μπορούν αυτέ να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε κατάρτιση και δανειοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένα εξατομικευμένα πλέον μέτρα τα οποία θα προωθήσουν την κατάσταση των γυναικών, να ενθαρρύνουμε τι γυναίκε κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργούν, να ιδρύουν επιχειρήσει χωρί να φοβούνται ότι θα διαταραχθεί η ισορροπία μεταξύ προσωπική και επαγγελματική ζωή. παρακαλώ. Thank you. Um, I... Ευχαριστώ στη σημερινή συζήτηση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα έχω μια ανανεωμένη αίσθηση του τι εστί εφικτό. Στη Βόρεια Ιρλανδία έχουμε μια νέα υπουργό. Αυτό είναι πρωτιά για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για το κόμμα μου. Γιατί έγινε εκείνη επικεφαλής του κόμματος. Είναι μια, ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσοι πιστεύουν ότι με ποσοστώσεις και με mainstreaming και με το ε, να δίδονται στις γυναίκες ευκαιρίες, ε, όσοι τα πιστεύουν αυτά σίγουρα δεν μπορούν να θεωρήσουν ότι η Βόρεια Ιρλανδία έχει σημειώσει, πρόοδο. Όμως έχουμε δείξει ικανότητα, στεναρή θέληση να επιτύχουμε και κυρίως δια της Υπουργού μας. Και γι' αυτό το, το μήνυμά μου είναι σαφές αυτή την έκθεση. Στηρίζω το στόχο σας να καταλύσετε κάθε είδους εμπόδιο άφηξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Ναι, θέλω την άρση των εμποδίων να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση. Ναι, θέλω οι γυναίκες να έχουν μια καλύτερη θέση στην κοινωνία και να μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρησιακές τους και επιχειρηματικές τους δεξιότητες, αλλά δεν συμφωνώ με την ιδέα των ποσοστώσεων. Άρκιν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι μια σημαντική έκθεση για την γυναική επιχειρηματικότητα και με χαρά την υπερψήφισα. Εάν δούμε τα νούμερα, καταλαβαίνουμε ότι το 31% ε, των επιχειρηματιών σε όλη την Ευρώπη είναι γυναίκες. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίξουμε τη γυναική επιχειρηματικότητα. Μία από τις δεξιότητες που έχουμε και μία από τις δυνατότητες είναι η μικροπίστωση, microfinance. Όμως ο λόγος γυναικών και ανδρών, ανδρών και γυναικών ήταν 60 προς 40. Ε, ε, για κάθε 60 άντρες που υπέβαλαν αίτηση, μόνο 40 άνδρες είχαν υποβάλει. για κάθε 60 άνδρες, μόνο 40 γυναίκες είχαν υποβάλει αίτηση. Θα πρέπει να έχουμε gender mainstreaming και στην κατανομή των κονδυλίων και νομίζω ότι τα νούμερα από τη μικροπίστωση αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα δίκτυο, ευρωπαϊκό δίκτυο, για την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Και χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει μια διαδικτυακή πλατφόρμα με κατάρτιση, με συμβουλές, με επιχειρηματικές δράσεις και θα έχουμε και γυναίκες επιχειρηματικούς αγγέλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περνάμε τώρα στην έκθεση Πλούρα Μπόιλαν. Παρακαλώ, πρώτος ο Απουσιάζει. Τζιτνάνσκα. Τζιτνάνσκα, τότε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πλούρα για αυτή την έκθεση. Ε, βλέπουμε πολλά θετικά στοιχεία στην έκθεση αυτή και πραγματικά είναι θετικό ρέθισμα για τις χώρες μέλη. Αυτό το οποίο εγώ θεωρώ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η έκθεση αυτή λαμβάνει υπόψη της ε, το θέμα της ότητας των ευκαιριών. Η έκθεση αυτή είναι μια έκκληση προς τις ε, αρμόδιες αρχές να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των ε, αναπήρων, ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν όλες οι ανισότητες. Η έκθεση αυτή επισημαίνει την ανάγκη της ε, περιεκτικής μάθησης αλλά και της χρηματικής στήριξης των αναπήρων. Θα ήθελα ε, να σας τονίσω το εξής. Για μένα η έκθεση αυτή είναι σημαντική γιατί το βασικό θέμα εδώ είναι η ευελιξία. Ευελιξία έναντι των φοιτητών ούτε ώστε να μπορέσουν εκείνοι να διαμορφώσουν τις σπουδέ τους έτσι που να μπορούν να σπουδάσουν αυτό που τους καθιστά ευτυχείς στη ζωή. Η κυρία Κλούν, σας ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή εστιάζει την προσοχή της στους νέους ανθρώπους και στις ε, πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η ανεργία είναι ψηλότερη σε ορισμένες ε, χώρες της Ευρώπης, αλλά το 95 ήταν επίσης πολύ ψηλά τα ποστά της ενεργείας, ήδη πριν από 20 χρόνια. Ε, και βρισκόμαστε άρα εναντί σοβαρών ε, προκλήσεων. Η ανάπτυξη σημαντικών ε, δεξιοτήτων είναι το θέμα αυτής της έκθεσης, καθώς και η κατάρτιση και εκπαίδευση ε, θα πρέπει να, γίνει, να υπάρχει συνεργασία με τους εργοδότες στον τομέα αυτό, ούτως για την απόκτηση των ε, βασικών ε, δεξιοτήτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο, μια νέα εστίαση ε, σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο ε, γιατί η ακαδημαϊκή μόρφωση δεν παρέχει στους νέους τις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συμβούλιο δεξιοτήτων ε, στο οποίο να συμμετέχουν ε, οι εργοδότες καθώς και οι εκπαιδευτές ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε την επαρκή, τον επαρκή εξοπλισμό των νέων με τις νέες δεξιότητες. Η κυρία Μορβά έχει το λόγο. Ναι, εγώ θα απόσχω στην ψηφοφορία γιατί ε, στο σημείο 1α και γ, δηλαδή ότι 4 έως 6 εκατομμύρια νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργοι, ε, και επίσης ε, εμφανίζονται κάποιοι αριθμοί για ανέργους ε, το ποσοστό των ανέργων μεταξύ 15 έως 25 είναι 7 εκατομμύρια. Ε, στο σημείο Γ λέει ότι οι νέοι πλήττονται ιδιαίτερα από το φαινόμενο της ενεργείας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, να πω το εξής. Θα πρέπει να καλέσουμε την κυρία Μέρκελ ε, και το επιτελείο της να μας πούν ε, γιατί ε, κάτω από τέτοιες ε, συνθήκες προσκαλούν ε, εκατομμύρια ανθρώπων από την Αφρική ενώ υπάρχουν τέτοια τεράστια ποσοστά ανεργίας στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο κύριος Κιούτσουκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σημαντική η έκθεση αυτή γιατί καλούμε να αντιμετωπίσουμε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές η ενεργεία των νέων σε ορισμένα κράτα-μέλη φτάνει ακόμα και το 50%. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε στους νέους αυτούς τις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να γίνουν και υπεύθυνοι πολίτες συμμετέχοντες σε μια δημοκρατική πλουραλιστική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η αγορά εργασία τροποποιείται πάρα πολύ γρήγορα. Και να καταφέρουμε να προβλέψουμε εμεί από τώρα τι μελλοντικέ δεξιότητε πολλέ φορέ είναι αδύνατο. Οι φοιτητέ λοιπόν θα πρέπει να έχουν μια ευρεία διαπαιδαγώγηση και κατάργηση. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να έχουμε μεταξύ κρατών μελών ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση, ιδίω όσον αφορά την εφαρμογή ενός συστήματος προειδοποίηση όσον αφορά την αλλαγή των συνθηκών στην αγορά εργασία. Θα πρέπει να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση των φοιτητών, θα πρέπει να έχουν καλύτερε δεξιότητε, γλωσσικέ και άλλε μαθησικέ δεξιότητε και θα πρέπει να καταφέρουν να περνάνε εύκολα και πιο ομαλά από το σχολείο στην αγορά εργασία. Γέλη, παρακαλώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, εγώ επεψήφισα αυτή την έκθεση και μάλιστα πολύ ενεργά. Ε, υποστήριξα την έκθεση αυτή γιατί δεν υπάρχει κανένα σημαντικότερο θέμα από αυτό δηλαδή την ε, ε, τον εξοπλισμό των νέων στο συνεσέλφου στην αγορά εργασία. Τα νούμερα για την ανεργία των νέων είναι καταστροφικά. Δεν μπορούμε συνεπώς να ονειρευόμαστε μια ειρηνική Ευρώπη κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Θα πρέπει να ληφθούν επιγόντως ε, μέτρα. Και η έκθεση καταδεικνύει ε, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη των χωρών μελών και των κυβερνήσεων. Δεν κατανοώ γιατί η Ουγγρική κυβέρνηση ή το ε, θέλει προτίθεται να καταστρέψει τον γρικό εκπαιδευτικό σύστημα και δεν καταλαβαίνω γιατί οι εκπρόσωποι του Γιώργη ε, του ακροδεξιού κόμματος ε, απήχαν και δεν υποστήριξαν την εν λόγω έκθεση. Προτείνω σε όλους να πάρουν το κείμενο αυτό σαν βάση και να θεωρήσουν το θέμα αυτό στο σημαντικότερο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παραθέσω δύο αριθμούς που είναι ενδεικτικοί της μέχρι τώρα αδυναμίας μας να δράσουμε στο φλέγον ζήτημα της απασχόλησης των νέων πέντε εκατομμύρια νέοι άνεργοι στην ευρώπη δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας. γιατί δεν παρέχουμε στους νέους τις δεξιότητες που τους λείπουν ώστε αυτές οι κενές θέσεις εργασίας να γίνουν άμεσα δουλειές με προοπτική; τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους πόρους για να βελτιώσουν τα προσόντα και τις δεξιότητες των νέων ανθρώπων που θέλουν να προχωρήσουν όμως είναι ότι προφανές σε μερικές χώρες η ψευτομαθητεία τείνει να γίνει συνήθεια πρέπει εδώ και τώρα να πιέσουμε τα κράτη μέλη και να ενεργοποιήσουν τα συστήματα εποπτείας και παρακολούθησης της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων ώστε η μαθητεία να εξελίσσεται άμεσα σε θέση εργασίας. ταυτόχρονα οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τη νεανική εξωστρεφή επιχειρηματικότητα με προώθηση των νέων επιχειρηματιών στο εράσμους αλλά και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. ξέρετε είναι βήματα μικρά απλά αλλά απαραίτητα και σε πολλά κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου χώρας προέλευσης της ελλάδος δεν έχουν γίνει επαρκώς. σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαμίκινς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή του κυρίου Πλούρα και ιδιαίτερα ευχαρίστω γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την ανική ανεργία μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες για την οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η δική μου μάλιστα τη χώρα, τη Λετωνία, η νεανική ανεργία αποτελεί πραγματική πληγή αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Οποιαδήποτε λοιπόν μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η οποία θα οδηγήσει σε μείωση αυτή της ανεργίας, οποιαδήποτε πολιτική θα μπορούσε να μειώσει αυτή την ανεργία είναι πραγματικά ευπρόσδεκτη. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι να συνειδητοποιήσουμε και το σε αυτό και η πρόταση αυτή, ότι όσοι βρίσκονται κάτω των 25 θα πρέπει να έχουν και τα απαραίτητα μέσα τα οποία θα παρέχονται από το κράτος προκειμένου να μπορούν τελικά να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και βέβαια η μείωση της ανεργίας θα πρέπει να γίνει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στις χώρες Αντολικής Ευρώπης. Ο κύριος Σόγκορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. 20% πάνω από 20% είναι η νεανική ενεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθο τη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στι χώρε μα. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει εμεί συνεχώ να δίνουμε μάχη προκειμένου το ζήτημα αυτό να συμπεριλαμβάνεται πάντα στα θέματα συζήτηση. Η έκθεση πολύ σωστά εντοπίζει το γεγονό τη έλλειψη δεξιοτήτων για τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από τα σημαντικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα κράτη-μέλη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι πολλές χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της πρώιμης αποχώρησης από το σχολείο. Έχουμε μεγάλα ποσοστά αποχώρηση από το σχολείο, εγκατάλειψη σχολείου σε κοινωνικές ομάδες όπως αυτές των Ρωμά. Νομίζω ότι στα πλαίσια των στρατηγικών απασχόληση Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να κεντρωθούμε περισσότερο στα ζητήματα αυτά, να επικεντρωθούμε στο εκπαιδευτικό σύστημα και να καταφέρουμε να κρατήσουμε όλο και περισσότερο παιδιά και νέου στο σχολικό σύστημα προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση έπειτα στην αγορά εργασία. Ο κύριο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι με χαρά μου στήριξα αυτή την έκθεση και ε, ψήφισα σύμφωνα με τις επιταγές της ε, πολιτικής μου ομάδας. Είναι κρίμα η κατάσταση με τους νέους ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικό κρίμα. Το είδα αυτό και στη δική μου χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Νέοι άνθρωποι, ε, πολλοί προσοντούχοι, να κάνουν αιτήσει για δουλειά, να πηγαίνουν για συνέντευξη και να λαμβάνουν πάντοτε την ίδια επιστολή. Με τα λύπης μου σας γνωρίζω ότι δεν καταφέρατε αυτή τη φορά να ε, πάρετε τη θέση εργασίας, ξαναπροσπαθήστε καλή τη σας τύχη. Και αυτή την επιστολή την έχουν λάβει επανειλημμένως οι νέοι. Απογοητεύονται και γι' αυτό είχαμε την τεράστια διαρροή εγκεφάλων στην Ιρλανδία έφυγαν κατά συρροή οι νέοι από τη χώρα. Ξέρω ότι η κατάσταση οικονομική της Ιρλανδίας βελτιώνεται. Θα έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 6% φέτος και επιστρέφουν νέοι για να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο και στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πόσπισιλ παρακαλώ. Ναι, εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση γιατί η ανεργία και η νεότητα και η απασχόληση είναι από τα, θα πρέπει να είναι από τα δυνατά σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, για να το πετύχουμε θα πρέπει να έχουμε μια ενεργό πολιτική και χαίρομαι πάρα πολύ που υποψηφίστηκε αυτή η έκθεση. Μια άλλη σύνδεση είναι εδώ στο θέμα της απασχόλησης των νέων είναι η κατάρτιση. Ε, ε, πολύ συχνά μια εκπαίδευση αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο δεν είναι Γι' αυτό θεωρώ ότι προγράμματα όπως είναι το Εράσμος και εγώ ιδίως ως πανεπιστημιακός καθηγητής γνωρίζω ότι αυτά τα προγράμματα βελτιώνουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις ε, ικανότητες αλλά επίσης δίνουν στους νέους την, την δυνατότητα να οριμάσουν εάν ζήσουν ένα-δύο χρόνια στο εξωτερικό. Ε, μου αρέσει επίσης το νέο πρόγραμμα Εράσμους για νέους επιχειρηματίες και εν γέννη θεωρώ πολύ θετική αυτή την έκθεση και χαίρομαι που εγκρίθηκε. Πετήρη παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή περιγράφει κάποια από τα πολύ βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι στι χώρε ευρωπαϊκής Ένωση και στην Κροατία. Σύμφωνα με δεδομένα τη Eurostat στην Κροατία, το ποσοστό ενεργείας για τους νέους κάτω την 25 το δεύτερο τρίμηνο του 2015 ανερχόταν στο 43,1%. Δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι η Κροατία βρίσκεται στην πρώτη θέση, στις πρώτες θέσεις τουλάχιστον, της νεανικής ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι τα μέτρα τα οποία προτείνονται στην έκθεση αυτά μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό λοιπόν τόσο τα κράτη-μέλη όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσουν πολιτικές που θα επιτρέψουν στους νέους να αποκτήσουν τις δεξιότητες αυτές που χρειάζονται για να γίνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Ως προς αυτό θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία αυτή του κυρίου Πλούρα, ο οποίο ζητά να έχουμε καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στι δημόσιε υπηρεσίε στην κοινωνία των πολιτών, τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις επιχειρήσεις. ο επιχειρηματικό τομέα. Θα μπορούσε και αυτό να αποφεληθεί και από του νέου, αλλά και το γεγονό ότι θα δημιουργηθούν κατά αυτόν τρόπο και νέε θέσει απασχόληση. Καλωσορίζω το ότι η έκθεση τονίζει μια διατομιακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ε, νεανικής ανεργίας. Ε, επίσης τονίζει την ανάγκη να έχουμε μια βάση δεδομένων ως προς τα προσόντα. Πράγματι, ε, τα προσόντα είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ των νέων και πρέπει να έχουμε καλή σύνδεση μεταξύ της διοίκησης των επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού συστήματος έτσι ώστε μια δραστηριότητα να γίνει πραγματική ευκαιρία. Το δίκτυο πρέπει να περιλαμβάνει επιχειρήσεις και κυρίως μικρομεσαίες, παρόχους εκπαίδευσης και να υπάρχουν βασικές σχέσεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την εθνική αρμοδιότητα. Ωστόσο, ο στόχος να έχουν μέλλον οι νέοι στην κοινωνία μας είναι σημαντικός και είναι αυτός που ε, τεκμηριώνει την ανάγκη υπερψήφισης της έκθεσης. Έχουμε και θελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με τους νέους. Στη Βόρεια Ιρλανδία η υλοποίηση αυτού του προγράμματος έχει προσκρούσει σε κολλήματα γραφειοκρατικά και σε διαφόρων ειδών ε, περιορισμούς. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια. Αυτό που μου αρέσει σε αυτή την έκθεση είναι που δίνει οι πρακτικές συμβουλές για να αντιμετωπίσουμε το θέμα με τους 7,5 εκατομμύρια νέους που δεν είναι ούτε σε εκπαίδευση, ούτε σε κατάρτιση, ούτε σε δουλειά. Βέβαια, πολύ συχνά έχουμε υπερβολικά πολλά προσόντα ή άλλοτε έχουμε ανεπαρκή προσόντα. Χρειαζόμαστε στέρεες εταιρικέ σχέσεις ε, μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κοινωνικών εταίρων και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να αφομοιώνονται και να ενσωματώνονται καλύτερα οι νέοι στην αγορά εργασίας. Και αυτό μπορεί να γίνει με την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας. Η έκθεση τονίζει ότι είναι σημαντικό να ταιριάξουμε τις δεξιότητες με τις δουλειές, αλλά πρέπει να έχουμε και μια συνολική παιδεία. Η, ε, εκπαιδεύεται κανείς, πηγαίνει σχολείο για να μάθει για τη ζωή, όχι μόνο για να μάθει για τη δουλειά και επίσης το να υπάρχει mentoring ε, έτσι ώστε να ε, πηγαίνουν ομαλά οι νέοι από το σχολείο στη δουλειά είναι μια ιδέα που αξίζει στήριξης. Υπάρχουν πολλές θέσεις απασχόλησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη χρήση παραδοσιακών δεξιοτήτων. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Κάλλας και Γκέπχαρτ. Ο κύριος Πόσπης είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Θεωρώ ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες της α, τρέχουσας εντολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν καταφέρουμε να αυξήσουμε τις ψηφιακές online πωλήσει και μάλιστα τις διασυνοριακές τέτοιες πωλήσει θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος. Έχουμε το χώρο Σέγγεν, υποτίθεται ότι δεν έχουμε σύνορα, αλλά δυστυχώ βλέπουμε ότι υπάρχουν σύνορα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτά πρέπει να καταρριφθούν. Οι μελέτε που έχουν λάβει η χώρα καταδεικνύουν ότι όλο και περισσότερε επιχειρήσει πουλούν αγαθά και υπηρεσίε εγχωρίω, αλλά δυστυχώ δυσκολεύονται πάρα πολύ να πουλήσουν αγαθά και υπηρεσίε διασυνοριακά. Στη χώρα μου είναι 26% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πουλούν υπηρεσίες και αγαθά επιγραμμικά, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφέρνει να παράσχει υπηρεσίες και αγαθά διασυνοριακά. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε τις επιγραμμικές διασυνοριακές πωλήσει. Μπενίτο Τζιλουάγκα, παρακαλώ. Nos hemos abstenido en la votación sobre el informe del mercado único digital. Ε, εμείς υπερψηφίσαμε την έκθεση αυτή για την ψηφιακή οικονομία και δεν ε, ε, θεωρούμε ότι μια ενιαία αγορά δεν είναι πάντοτε η λύση, ούτε ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να δημιουργήσει θέσει απασχόληση ψηλή ποιότητα. Η έκθεση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να ευνοήσει περισσότερο τι μεγάλες επιχειρήσει. Εμείς έχουμε καθέσει τροπολογίες ούτε ώστε η οικονομία τη αγορά, να ε, περιλαμβάνει και κοινωνική προστασία. Επιθυμούμε να πάμε, να πάει μακρύτερα η Επιτροπή όσον αφορά την ουδετερότητα του διαδικτύου το ίντερνετ θα πρέπει να είναι ένα συνολικό χώρος για την επικοινωνία και τον δημοκρατικό μετασχηματισμό, όπως για παράδειγμα συνέβη στην ε, Αραβική Άνοιξη. Το ίντερνετ δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα νέο εμπορικό προϊόν, εμπορικό χώρο. Ε, Η κυρία Μορβάη, παρακαλώ. όσον αφορά την ε, ψηφιακή αγορά υπερψήφισα την έκθεση αλλά θεωρώ ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι 4% μόνο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάνει πωλήσει online μέσω της χρήσης του ίντερνετ. Μεταξύ αυτών είναι ιδιαίτερες μικρές επιχειρήσεις. Ε, και ξέρω τι γίνεται ε, σε διάφορα νοικοκυριά όπου μικρά παιδιά έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ ή και ηλικιωμένοι. Υπάρχουν επίσης ε, άνθρωποι οι οποίοι παράγουν στο σπίτι τους μαρμελάδες ή άλλα τοπικά προϊόντα και θα ήταν πολύ σημαντικό να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους αυτά μέσω του ίντερνετ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, όταν ψέψω την πατρίδα μου θα ρωτήσω τις αρχές να με ενημερώσουν, να δω τι γίνεται με αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και να μου πούν σε ποιο βαθμό είναι δυνατές οι πωλήσει online για αυτές τις πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Γιατί ε, πραγματικά θα με χαροποιούσε αυτό ιδιαίτερα. Η κυρία Μπόρτσαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όλοι θα πρέπει να τηρήσουμε τους πολύ αυστηρούς κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και την περίοδο αυτή των 14 ημερών που προβλέπεται στην έκθεση αυτή. Αυτό είναι σωστό, αλλά τελικά επιβαρύνει οικονομικά τις επιχειρήσεις και υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι φοβούνται να κάνουν ψηφιακές αγορές στο ίντερνετ γιατί θεωρούν ότι ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να καθορίσουμε τελικά αν όντως ο πολιτής είναι κατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βάλουμε ένα ειδικό σήμα εμπιστοσύνης θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για όλους. Τώρα το ζήτημα των παραδόσεων επίσης των προϊόντων και αυτό είναι πολύ σημαντικό και εκεί πέρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και μικρότερο κόστος. Δεν μπορούμε ποτέ να περιμένουμε ότι θα διευρυνθούν, ότι θα επεκταθούν αυτές οι επιγραμμικές πωλήσει αν κοστίζει πάρα πολύ σημαντικά το σύστημα αυτό των προϊόντων. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Μίτση, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Συντοποιούμε πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά. Η νέα αυτή ψηφιακή επανάσταση δίνει πάρα πολλέ δυνατότητε προκειμένου να καταφέρουμε να κοινοτομήσουμε σε πάρα πολλού τομεί τη ευρωπαϊκή οικονομία και να αλλάξουμε την ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η ολοκλήρωση λοιπόν τη ψηφιακή ενιαία αγορά και το να γίνει αυτή προσβάσιμη σε όλου του πολίτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα θα δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πολίτε, οι καταναλωτέ και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και όσοι ανήκουν σε ευάλωτε ομάδε να μπορούν να προστατεύονται καταλληλώ και να έχουν ε, τη δυνατότητα να κάνουν ε, προσφυγέ, δικαστικέ προσφυγέ όσον αφορά αυτέ τι ψηφιακέ υπηρεσίε. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δώσουμε στου πολίτε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ευφυεί τεχνολογίε προκειμένου να αποφεληθούν περισσότερο από τι ψηφιακέ αυτέ υπηρεσίε. Θα πρέπει οι επιχειρήσει να προετοιμαστούν όλο και περισσότερο για τη νέα ψηφιακή εποχή για να ανταποκριθούν στι ανάγκε του μέλλοντο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καπούτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κείμενο το οποίο ψηφίσαμε διευκρινίζει με απόλυτη ακρίβεια ποιε είναι οι ευκαιρίε και οι προκλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια μια μελλοντική ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να συνειδητοποιήσει ποια είναι τα διδάγματα τη έκθεση αυτή. Ζητάμε όλο και περισσότερο τη δυνατότητα διασυνοριακών πωλήσεων οι οποίε είναι ιδιαίτερα περιορισμένε αυτή τη στιγμή. Επίση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιβληθούν συγκεκριμένοι ενοποιημένοι κανόνε για το copyright και τα δικαιώματα του δημιουργού και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούν όλοι οι δημιουργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να αποφεληθούν από τα έργα τα οποία πολλούνται στην ε, ψηφιακή αγορά. Να καταπολεμήσουμε επίση την πειρατεία και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι ο ρόλο των μεσολαβητών και των ε, online πλατφόρμων. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει την απαραίτητη σημασία που δίνεται από τις νέες τεχνολογίες, τις τεχνολογίες big data, από το cloud computing, καθώς επίσης και από πολλές άλλες τεχνολογίες. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, αν αποφεληθούμε από τις νέες αυτές τεχνολογίες, θα δημιουργήσουμε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για τους νέους μας. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και πάλι υπερψήφισα αυτή την έκθεση και ακολούθησα τις ε, πολιτικές επιταγές της πολιτικής μου ομάδας. Είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Σχετίζεται με όλα τα άλλα θέματα που συζητήσαμε, την ανεργία των νέων για παράδειγμα, την γυναική επιχειρηματικότητα επίσης. Είναι καταπληκτική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλές δουλειές, θέσεις εργασίας, χωρίς παραπάνω δαπάνε. 450 δις ευρώ μπορούν να υπάρξουν για την ευρωπαϊκή οικονομία εάν το καταφέρουμε να το κάνουμε σωστά. Και αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε σωστά. Και θα πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια στους επιχειρηματίες να είναι ευκολότερο οι άνθρωποι να πολλούν και να αγοράζουν στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ ο κύριος Χάρκιν. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με χαρά στήριξα αυτή την έκθεση για την ενιαία ψηφιακή αγορά, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πλαίσιο για το κοινό ψηφιακό μας μέλλον. Δεν στήριξα την τροπολογία 24, γιατί αυτή η τροπολογία προσπαθεί να φέρει κάποια ισορροπία και καλώς αναγνωρίζει από τη μία ότι η ψηφιοποίηση οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτονομία και σε ευελιξία από την άλλη πλευρά οδηγεί σε νέες προκλήσεις όπως είναι η παράταση του ωραρίου εργασίας η τεράστια κόπωση εργασιακή και ούτω καθεξής την ε, καταψήφισα για τη από την Επιτροπή να μελετήσει ε, τα spillover effects, τα αποτελέσματα από την ψηφιοποίηση σε άλλους τομείς όπως είναι για παράδειγμα η ανάπτυξη των γνωσιακών δεξιοτήτων των παιδιών και δεν το έκανε. Ναι, καλό είναι το ψηφιακό και όλοι θέλουμε να είμαστε όλο και πιο ψηφιακοί και ψηφιοποιημένοι, αλλά δεν μελετούμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Η ψηφιακή αγορά δεν είναι από μόνη της επεργετική ή ε, καταδικαστική. Πρέπει να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά, να οξύνουμε τα θετικά και να ελεγχιστοποιήσουμε τα αρνητικά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνονται έτσι οι αιτιολογήσεις ψήφου και διακόπτη συνεδρίαση μέχρι τις 3.